των ηρημένων συναδέλφων. Η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων αντιμετώπισε το θέμα της εφαρμογής του άρθρου 47 του κανονισμού. Βάσει του άρθρου 201, παράγραφος 3, προτείνει την εξή διατύπωση για το άρθρο αυτό. Και παραθέτω. Στα πλαίσια της εξέτασης μιας διεθνούς συμφωνίας βάσει του άρθρου 83 του κανονισμού, η διαδικασία με συμμετοχή περαιτέρω επιτροπών βάσει του άρθρου 47 δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή της ενισχυμένη συνεργασία των Επιτροπών βάσει του άρθρου 75. Αυτή η διατύπωση θεωρείται ως ε, ηλυμένη όταν δεν υπάρξουν, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις σε σχέση με την έγκριση των πρακτικών συνεδριασή μας. Η τελευταία ανακοίνωση, η αρμόδια επιτροπή μου έχει μεταφέρει μία έκθεση σε σχέση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου